θα επαναληφθεί αύριο το πρωί και υπάρχει η περίσσια διάταξη στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και τους κυρίου